Καλησπέρα σας. Έχουμε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι η συμφωνία ανάμεσα σε Καναδά και Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την επεξεργασία του PNR. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε την άποψη της ε, νομικής υπηρεσίας για την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου της 26ης Ιουλίου που αφορά στη συμφωνία ανάμεσα σε Καναδά και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα σχετικά με το θέμα μας. Ε, αυτά έγιναν μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε με βάση το 218 11. Θα ακούσουμε λοιπόν η νομική υπηρεσία και βεβαίως μετά θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να τοποθετηθούν. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. The European Parliament decided On the 24th of November 2000... Στη νομική υπηρεσία. Όπως αποφασίστηκε λοιπόν, ε, μάλλον όπως είπατε, είχε ζητηθεί η άποψη της νομικής υπηρεσίας για δύο θέματα. Το πρώτο ερώτημα ήταν η συμβατότητα της ε, Διεθνούς Συμφωνίας ε, αυτή του Καναδά με την συμφωνία για το PNR. Βέβαια, αυτά έχουν άμεση σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, κυρίως με το ε, δικαίωμα της ιδιωτικής σφαίρας και της πρόσβασης στα δεδομένα. Το δεύτερο θέμα ήταν η επιλογή της νομικής βάσης. Το Συμβούλιο είχε προτείνει να ε, εγκριθεί η συμφωνία με βάση το άρθρα 82 και 87 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρόκειται για την ε, συνεργασία σε θέματα εγκληματικής φύσεως. Τώρα, το θέμα είναι κατά πόσον πράγματι με βάση το 16 υπάρχει η σωστή νομική βάση. Εκεί υπάρχει η νομοθεσία για την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων. Αυτά το 16 Τώρα, στις 26 Ιουλίου του 2017 ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τοποθετήθηκε, αποφάνθηκε τελεσίδικα ε, από αυτών των δύο θεμάτων και έχουμε πλέον όπως σας είπα την ε, τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφαίνεται όσον αφορά στη συμβατότητα μιας διεθνούς συμφωνίας με το χάρτη. Αυτό είναι κάτι το καινούριο, καινοφανές. Και μάλιστα η απαντήσει του Ευρωδικαστηρίου είναι πολύ λεπτομερεί. Εγώ θα τι παρουσιάσω συνοπτικά. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξή. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα για τη νομική βάση, το δικαστήριο δηλώνει ότι η νομική βάση που προτίθηκε αρχικά από το Συμβούλιο δεν είναι σωστή. Αντί για τα 82 και 87, η νομική βάση θα έπρεπε να βασίζεται στα άρθρα 16 και 87. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι το δικαστήριο δηλώνει ότι η διεθνή Συμφωνία δεν συμβαδίζει πλήρως με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τουλάχιστον στην κείμενη μορφή του. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια τμήματα της συμφωνίας συμφωνούν με το χάρτη, όχι όλα, κάποια, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα που ε, δεν συμμορφώνονται. Και θα ήθελα να εξηγήσω δύο θέματα. Όσον αφορά στη νομική βάση, θα είμαι σύντομος, όπως σας είπα, η νομική βάση προτινόμενη είναι ε, δικαστική συνεργασία σε θέματα εγκλημακής φύσεως με βάση τα άρθρα 82 και 87 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαστήριο είπε ότι το 82 για τη δικαστική συνεργασία δεν ισχύει, διότι οι διεθνείς ε, συμφωνίες δεν πρέπει να ασχολούνται με τη δικαστική συνεργασία, άρα αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί. Βέβαια το δικαστήριο λέει το 87 για την τη συνεργασία αστυνομικών αρχών. Εκεί ε, η συμφωνία έχει σχέση με τη συνεργασία, αλλά το δικαστήριο λέει επίσης ότι το άρθρο 16 της συνθήκης που αφορά την προστασία των δεδομένων και αυτό ε, είναι αδιάφορο, γιατί ένας από τους στόχους της συμφωνίας είναι να διασφαλιστεί η προστασία δεδομένων και ε, ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα. Ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες για νομική βάση. Αφενός, συνεργασία νομικών αρχών, αφετέρου, ε, προστασία εντομένων, ποια είναι η κατάλληλη νομική βάση που πρέπει να ισχύει. Εδώ λοιπόν το δικαστήριο μπαίνει στο περιεχόμενο της συμφωνίας και καταλήγει στο ότι και οι δύο πτυχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Δεν μπορεί να τις διαχωρίσει το δικαστήριο, άρα και το 16 και το πρέπει από κοινού να αποτελούν νομική βάση. Εδώ έχουμε διπλή νομική βάση, 16 και 87. Αυτό είναι εξαίρεση, για τις γενικές γραμμές με βάση την ε, ε, τρέχουσα νομολογία δεν ήθιστε κάτι τέτοιο, αλλά όπως λέει το δικαστήριο, η διαδικασία για την θέσπιση των πράξεων της νομικής βάσης, η διαδικασία πρέπει να είναι συμβατή. Και εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε το άρθρο 87 πέφτει, εμπίπτει στο κεφάλαιο υπαριθμών 5 και Εκεί τα, ισχύουν τα πρωτόκολλα για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Δανία, την Ιρλανδία. Άρα εδώ υπάρχει κάποιο θέμα και το δικαστήριο εξηγεί στην γνωμοδότησή του ότι για αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι η συμφωνία δεν ισχύει πουδενή για τη Δανία λόγω της κατάστασης της Δανίας και όσον αφορά Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία και οι δύο προαιρετικά προσεχώρησαν στη συμφωνία. Άρα δηλαδή κάτω από αυτές τις ειδικέ συνθήκες, το δικαστήριο λέει ότι είναι δυνατόν να εφαρμόζονται το 16 και το 87 από κοινού. Γι' αυτό έχουμε λοιπόν ε, διπλή νομική βάση. Πάω τώρα στο άλλο ερώτημα που αφορά στο χάρτη, αν υπάρχει συμμόρφωση με το χάρτη. Σας είπα, είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο στην τελεσίδικη απόφασή του εξετάζει ένα τέτοιο θέμα. Αρχικά το δικαστήριο ε, διαβεβαιώνει ότι πράγματι ο χάρτης ισχύει οποτεδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει διεθνείς συμφωνίες. Άρα δεν πρόκειται ε, για ένα χάρτη που είναι εσωτερική ε, νομοθεσία. Ο χάρτης ισχύει για όλες τις ενωσιακές πράξεις και τις διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται. πρέπει κανείς να διορτηθεί κατά πόσον κάθε φορά αυτές οι διεθνείς συμφωνίες είναι συμβατές με το χάρτη. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο το δικαστήριο αναλύει πώς ισχύει ο χάρτης. Γιατί κατ' ουσίαν το δικαστήριο ε, εφαρμόζει την ίδια μέθοδο στην εφαρμογή του χάρτη, όπως και όταν πρόκειται για ενωσιακή νομοθεσία. Δεν πρόκειται κάτι το ιδιαίτερο, άρα δηλαδή ε, πρόκειται για τις ίδιες αρχές, ε, για την ίδια μέθοδο ανάλυσης, ε, για το κατά πόσον ισχύουν οι αρχές του χάρτη. Αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν οι λεπτομέρειες αυτής της συγκεκριμένης συμφωνίας. Και όσον αφορά αυτό το θέμα, τη μέθοδο εφαρμογής, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω Αυτά που έχουν ήδη αποφασιστεί από το δικαστήριο σε προηγούμενη απόφαση το 14, τον Απρίλιο του 2014 για την Ιρλανδία. Όπως ξέρετε, πρόκειτο για την οδηγία σχετικά με την ε, ε, διαφύλαξη των δεδομένων και το δικαστήριο είπε ότι ε, η απόφαση δεν ισχύει γιατί δεν συμβατεί με το χάρτη. Και έγινε κάποια συζήτηση για το πώς αυτή η απόφαση θα μπορούσε να ισχύει και για άλλους τομείς. Και η νομική υπηρεσία τοποθετήθηκε, εκλήθη να τοποθετηθεί. Προτείναμε λοιπόν ότι το αιτιολογικό το δικαστήριο από προηγούμενη απόφαση μπορεί να ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις. Ε, το ίδιο λοιπόν ε, σκεπτικό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το δικαστήριο μας δείχνει πώς ε, αυτό το σκεπτικό μπορεί να ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις. Είπαμε ότι ισχύει το ίδιο σκεπτικό και σε άλλες περιπτώσεις. Το δικαστήριο αποφάσισε για τα ψηφιακά δικαιώματα της Ιρλανδίας. Έχουμε την τελευταία απόφαση τελετού και έτσι αυτή η γνωμοδότηση επιβεβαιώνει την προσέγγιση του δικαστηρίου. Δεν πρόκειται μόνο για την ε, διαφύλαξη των δεδομένων, αλλά γενικότερα. Όπως σας είπα, δεν σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις καταλήγουμε σε δύο αποτέλεσμα, αλλά τώρα έχουμε κάποιες ε, κατευθύνσεις για την ε, γενικότερη προσέγγιση. Η προσέγγιση του δικαστηρίου είναι σε τρεις φάσεις. Πρώτα ε, διερωτάτε κατά πόσον ισχύουν κάποια άρθρα του χάρτη. Αν κάποια άρθρα και κάποια δικαιώματα ισχύουν, το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον παραβιάζονται αυτά τα δικαιώματα. Και αν υπάρχει αυτό, το δικαστήριο διερωτάται πόσο σημαντική είναι η παραβίαση. Αν είναι σημαντική η παραβίαση, μετά το δικαστήριο αναλύει πολύ προσεκτικά κατά πόσον αιτιολογείται η παραβίαση ή όχι. Το δικαστήριο εξετάζει πολύ προσεκτικά την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας και εδώ ακολουθεί την ίδια προσέγγιση, τις τα ίδια βήματα. Το βασικότερο ε, είναι το τελευταίο που αφορά στην αναγκαιότητα και την αναλογικότητα. Εκεί το δικαστήριο με λεπτομέρειες ε, εξηγεί ε, το περιεχόμενο των διεθνών συμφωνιών και εξηγεί επίσης ε, το ότι κάθε τμήμα των διεθνών συμφωνιών ε, συμβαδίζει με τις αρχές και πρέπει να συμβαδίζει με τις αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Και καταλήγει ότι ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν συμβαδίζουν με το χάρτη. Για να κατανοήσει κανείς πώς γίνονται όλα αυτά το δικαστήριο, χωρίζει όλο αυτό σε τρεις φάσεις και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει το να τα εξτάσει κανείς ε, με κάποια σειρά. Οι τρεις αυτές φάσεις που εφαρμόζει το δικαστήριο είναι ένα ταξίδι που κάνει ένας επιβάτης προς τον Καναδά, μένει στον Καναδά, στην πρώτη φάση είναι όταν ο επιβάτης μπαίνει στο αεροπλάνο, πετάει προς Καναδά, φτάνει στον Καναδά και περνάει μέσα από συνοριακό έλεγχο. Αυτή είναι η πρώτη φάση, η πρώτη μέρα, διαρκεί κάποιες ώρες. Η δεύτερη φάση κατόπιν είναι κατά τη διάρκεια της παραμονής του επιβάτη στον Καναδά, λίγες μέρες, λίγοι μήνες ενδεχομένως. Ε, μικρή η περίοδος, σύντομη. Η τρίτη φάση είναι μετά την, ε, από τότε που φεύγει ο επιβάτης. Το δικαστήριο λοιπόν εξτάζει αυτές τις φάσεις και διερωτάται. Δικαιολογείται η παρέμβαση μέσω του συστήματος PNR. Στην πρώτη φάση, πριν λοιπόν ο επιβάτης ε, του επιτραπεί να μπει στον Καναδά, εκεί το δικαστήριο δέχεται ότι το σύστημα PNR δικαιολογείται και ότι η διαβίβαση όλων των στοιχείων επιβατών σε μια τρίτη χώρα μπορεί να είναι αποδεκτή και η χώρα αυτή μπορεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα. Σας λέω όμως ότι αυτό αφορά στην πρώτη φάση, όταν δηλαδή το αεροπλάνο ταξιδεύει προς Καναδά. Και έτσι οι αρχές του Καναδά έχουν το δικαίωμα πριν κάποιος φτάσει να μπορούν να εξετάσουν αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ασφάλειας. Και ο λόγος που τα δέχεται όλα αυτά είναι ότι με βάση το διεθνές δίκαιο όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε ελέγχους ε, σε σχέση με τους επιβάτες ε, που φτάνουν στο έδαφος τους. Άρα δηλαδή ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μεταφέρονται τα δεδομένα ενός επιβάτη προς μια τρίτη χώρα, έτσι ώστε αυτή η τρίτη χώρα να εξετάζει τους επιβάτες την ώρα που αφήκνυνται. Ως εκ τούτου το σύστημα PNR μπορεί να εφαρμόζεται σε αυτή την πρώτη φάση. Με δύο όμως βασικές προϋποθέσεις που ξεκαθαρίζει το δικαστήριο. Πρώτον, δεν μεταβιβάζονται ευαίσθητα δεδομένα. Δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για τη διαβίβαση των ευαίσθητων δεδομένων και η δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι το δικαστήριο εξηγεί πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα επεξεργασίας στοιχείων PNR. Γίνεται επεξεργασία όλων των δεδομένων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό είναι αποδεκτό, γιατί είναι ένας τρόπος ε, ε, να γνωρίζει κανείς ε, ότι ένας επιβάτης δεν αποτελεί κίνδυνο, ότι υπάρχουν επιβάτες που ποτέ δεν έχουν διαπράξει κανένα δίκημα. Ως εκ τούτου, το PNR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστούν άγνωστοι ύποπτοι. Και ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να επεξεργαστούν ε, οι αρχές τα στοιχεία όλων των ε, επιβατών. Βέβαια, το δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι το σύστημα PNR είναι ένα σύστημα με βάση συγκεκριμένες παραδοχές. Παράλληλα, λέει το δικαστήριο ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι σε αυτή τη μέθοδο του profiling στις παραδοχές που είπαμε προηγουμένως. Οι παραδοχές αυτές, το προφίλ τέλο πάντων δεν θα πρέπει να, έχει, να είναι να περιλαμβάνει στοιχεία διακριτικής μεταχείρισης, ε, να μπορεί κανείς να αναθεωρήσει επίσης τους αλγορίθμους μέσα στο σύστημα που καταρτίζει το προφίλ, κάποιες μέθοδοι δηλαδή με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Καναδά ελέγχουν πώς γίνεται ε, η σύνταξη του προφίλ του επιβάτη. Και πρέπει να γίνονται και κάποιε συζητήσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά για να μην υπάρχουν διακρίσει στην ε, σύνταξη προφίλ του επιβάτη. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Δηλαδή ε, η νομολογία δεν περιλαμβάνει ούτε θέματα προφίλ, ούτε αλγορίθμους. Είναι κάτι καινούριο. Αυτό μπορούμε να το διαπραγματευτούμε με τον Καναδά και Τώρα πλέον το δικαστήριο λέει ότι όλα αυτά θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Αυτά μπορεί στο μέλλον να είναι σημαντικά. Αυτή είναι η πρώτη φάση, πριν φτάσει ο επιβάτης ε, στον ε, ε, έλεγχο διαβατηρίων. Η δεύτερη φάση, ο επιβάτη έχει περάσει από τον έλεγχο και μπορεί να μπει πλέον στον πενατά. Υπάρχουν δύο δυνατότητε, είτε κατά τη διάρκεια τη πτήση ε, γίνεται σημαντικό έλεγχο του PNR, ο οποίο και δεν αποκάλυψε κίνδυνο για κάποιο ιδιαίτερο επιβάτη, άρα επιτρέπεται η ε, ελεύθερη είσοδο, είτε το σύστημα PNR εντόπισε ως ενδεχόμενο κίνδυνο κάποιον επιβάτη και έτσι λοιπόν να τον υποδέχονται οι κοινωνικέ αρχέ στην άφηξη του Ωστόσο, στην ε, περίπτωση αυτή, μετά από ανάκριση του επιβάτη, διαπιστώνουν οι αρχέ, ε, ότι δεν υπάρχει κίνδυνο και άρα επιτρέπεται η είσοδο του. Και σε δύο περιπτώσει, λοιπόν, επιτρέπεται η είσοδο. Εδώ, λοιπόν, έρθει με διαφορετική οι συνθήκες. Αλλάζουν τα πράγματα. Επιτρέπεται η είσοδο του επιβάτη και η παραμονή του στον Καναδά για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλάζει, λοιπόν, η κατάσταση και είναι σημαντική η αλλαγή αυτή. Γιατί το δικαστήριο δεν αποδέχεται πλέον ότι θα πρέπει να υπάρχει συστηματικό καθορισμός του profiling των επιβατών, αυτό που γινόταν, αλλά δεν ζητά αυτόματα διαγραφή των δεδομένων σε αυτή τη φάση. Αποδέχεται το δικαστήριο ότι οι καναδικές αρχέ μπορούν να διατηρήσουν τα στοιχεία για τη διάρκεια τη παραμονή του επιβάτη στον Καναδά. Αλλά οι καναδικέ αρχέ δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά άμεσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το δικαστήριο επιμένει πρωτού υπάρχει στη δεύτερη φάση πρόσβαση από τι κοινωνικέ αρχέ στα δεδομένα. Θα πρέπει να στραφούν στο δικαστήριο και να ζητήσουν μια δικαστική έγκριση. Μόνο μετά από τη δικαστική έγκριση λοιπόν αυτοί έχουν πρόσβαση. Σημαντική αυτή η ασφαλιστική δικλίδα σε ό,τι αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια και την προσαγωγή των απαραίτητων αποδεκτικών στοιχείων. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και μοιάζει πλέον στην κατάσταση που έχουμε την διατηρήση των δεδομένων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με τα δύο συστήματα, το PNR, δηλαδή μετά την είσοδο του επιβάτη στη χώρα. Μπορούν να τεθούν τα στοιχεία αυτά, αλλά όχι να υπάρχει πρόσβαση χωρίς δικαστική απόφαση. Δεν είναι το PNR λοιπόν όπως γνωρίζουμε στην παρούσα φάση αυτό. Επίσης, οι άλλες κρατικές αρχές μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά PNR, όχι μόνο οι αρχέ φύλαξη των συνόρων, αλλά και πάλι θα πρέπει να υπάρχει δικαστική έγκριση και οι τρίτε χώρε επίση μπορεί να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά τα οποία αποθηκεύονται στον Καναδά στη διάρκεια αυτή, αλλά και πάλι οι τρίτε χώρε και αυτέ θα χρειαστούν έγκριση από τα δικά του δικαστήρια, τα εθνικά του δικαστήρια, πρώτου έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Και υπάρχει λοιπόν αυτή η επιπλέον ασφαλιστική δίκλυδα σε ό,τι αφορά τι τρίτε χώρε το δικαστήριο ζητά σχετική απόφαση και της ε, ε, Επιτροπής, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει διεθνή συμφωνία με τη χώρα αυτή που να επιτρέπει τη μεταφορά των δεδομένων και στις δύο περιπτώσεις αυτές μπορεί οι καναδικές αρχές να χορηγήσουν τα στοιχεία αυτά στις τρίτες χώρες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η μεταφορά των δεδομένων αυτών. Αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο. Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο είναι όταν ο επιβάτης φεύγει από τη χώρα, φεύγει από τον Καναδά. Ε, το δικαστηρίο θεωρεί ότι η κατάσταση τροποποιείται και πάλι. Γιατί σημειώνονται ότι ο επιβάτης θα πρέπει να ελεγχθεί όταν κατά την άφηξη του και υπάρχει δυνατότητα με δικαστική απόφαση να γίνει έλεγχο και στην παραμονή του, κατά την παραμονή του και όταν φεύγει πλέον ο επιβάτης από τον Καναδά, ουσιαστικά το δικαστήριο θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον ε, κίνδυνος ο οποίος να δικαιολογεί τη διατήρηση των δεδομένων. Άρα, όταν ο επιβάτης ε, αποχωρεί από τον Καναδά μετά από κάποιες ημέρες ή εβδομάδες, το δικαστήριο ουσιαστικά επί της αρχής απαιτεί διαγραφή των δεδομένων. Αυτό αποτελεί μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την υφιστάμενη προβλεπόμενη διαδικασία, όπου τα δεδομένα ουσιαστικά φυλάσσονται για πέντε έτη. Αυτή είναι η αρχή γιατί τη διαγραφή δηλαδή των δεδομένων των πιο πολλών επιβατών όταν αποχωρούν από τη χώρα. Ωστόσο, το δικαστήριο αποδέχεται σε κάποιε περιπτώσει κατά εξαίρεση, κατά εξαίρεση να μπορούν οι Καναδοί να διατηρούν τα δεδομένα για μεγαλύτερη περίοδο, μέχρι και πέντε χρόνια, αν σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια συντρέχουν λόγοι που α, μας κάνουν να πιστεύουν ότι αποτελεί κίνδυνο το συγκεκριμένο άτομο. Αυτό όμως αφορά με μερισμένο αριθμό επιβατών περιορισμένο αριθμό ατόμων των οποίων τα δεδομένα ε, διατηρούνται για πέντε χρόνια. Στοχευμένη διατήρηση λοιπόν δεδομένων κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό αποτελεί ένα παραλληλισμό, αν θέλετε, με τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά και τι σχετικέ ρυθμίσει. Όπω βλέπετε λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα τρία αυτά επίπεδα, είναι μεγάλε οι αλλαγέ σε σχέση με το εφιστάμενο μοντέλο PNR και ε, την ε, σταδιακή μείωση των περιορισμών των δεδομένων που μπορούν να διατηρηθούν και για το, ε, την περίοδο ρύθμιση τους και για την δυνατότητα πρόσβασης από πλευρά των αρχών στα δεδομένα αυτά. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί μια καλή σύνοψη του τι σημαίνει και τι προβλέπει αυτή η νέα συμφωνία. Άρα το σύστημα αποφανθεί το δικαστήριο το οποίο το, τρέχον σύστημα αποφανθεί το δικαστήριο ότι είναι παράνομο και θα πρέπει να αλλάξουν οι σημαντικέ διτάξει για να καταστεί σύνομο. Και επίση άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και το δικαστήριο, για παράδειγμα, απαιτεί οι επιβάτε του δεύτερου και του τρίτο επίπεδου αν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα με δικαστική απόφαση, θα πρέπει ενημερώνονται σε μετέπειτα χρονική στιγμή ο επίβατη για να ελέγχει κατά πόσο ήταν πραγματικά νόμιμη η πρόσβαση στα δεδομένα του. Και αυτό λοιπόν προβλέπεται. Και για να ολοκληρώσουμε, ποιε είναι οι συνέπειε ε, στη συμφωνία με τον Καναδά σύμφωνα με το άρθρο 218 της συνθήκης όταν το δικαστήριο ε, εκδίδει αρνητική συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί η Διεθνή Συμφωνία. Προφανώ τρέχουν οι λόγοι στην προκειμένη περίπτωση και τουλάχιστον η προκειμένη συμφωνία δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Φυσικά αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα εντολή του Συμβουλίου είναι να κάνει εκ νέου διαπραγμάτευση τη συμφωνία προκειμένου να συνάδει με, το, με τη χάρτα. Αλλά φαντάζομαι ότι γι' αυτό θα μα ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα φάση. Δεν χρειάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να γιατί πολύ απλά η συνθήκη ορίζει ότι δεν μπορεί να τέτοιες σε εφαρμογή συμφωνία και αυτό εξακολουθεί φυσικά να προβλέπει την δυνατότητα παρακολούθηση τη κατάσταση από πλευρά του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο φυσικά θα ενημερώνεται σε όλε τι φάσει των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Να είμαι βέβαιο ότι θα έχετε πάρα πολλέ ερωτήσει, αλλά ε, με χαρά να σα ε, απαντήσω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, να ακούσουμε τον εισηγητή πρώτα και μετά του συντονιστέ. Σοφή. Yes, thank you and... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμός και την νομική υπηρεσία για την διεξοδική αυτή ανάλυση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση. Που μας δίνει ας πούμε κάποιες δυνατότητες για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις και συμφωνίες. Το πρώτο που ήθελα να καταλάβω είναι τι έπεται. Και κατάλαβα ότι απλώς θα επανέλθει στο Συμβούλιο και την Κομισιόν. Αυτό και επομένω εμείς μπορούμε να διηγηθούμε στο ψήφισμά μας. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, τι επιπτώσει μπορεί να έχει αυτή η απόφαση για άλλου είδους συμφωνίες ή ακόμα και για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί Εξετάζοντας τα επιχειρήματα του δικαστηρίου, το PNR με τις ΗΠΑ ούτε από μακριά δεν πλησιάζει. Με την Αυστραλία ίσως είναι πιο κοντά, αλλά και εκεί υπάρχουν διαφορές. Και υπάρχει και η οδηγία. Επομένως, τι θα γίνει με όλα αυτά. πρέπει να συμπεράνουμε ότι αυτές οι άλλες συμφωνίες δεν θα εξεταστούν το δικαστήριο. Καλύπτουν τα κριτήρια, συμμορφούνται. Κάποιος πρέπει να διαβουλευθεί με το δικαστήριο. Θα γίνει αυτό από το ίδιο το δικαστήριο. Ποιος θα μας βεβαιώσει ότι ευθυγραμμίζονται με το χάρτη μελιωδών δικαιωμάτων ή ότι έχουν την κατάλληλη βάση, τουλάχιστον ως προς το άρθρο 16. Δηλαδή, τουλάχιστον επί του συγκεκριμένου στοιχείου, οι άλλες συμφωνίες έχουν εντύπωση ότι δεν συμμορφούνται. Επίσης το δικαστήριο λέει ότι η μαζική αποθήκευση δεδομένων όλων των επιβατών είναι κάτι που μπορεί να γίνει αλλά το δικαστήριο θεωρεί ότι αυτό επιτρέπεται επειδή είναι τμήμα διεθνού συμφωνίας, το οποίο θα υπονοούσε ότι δεν θα επιτρέπεται αν ήταν για ευρωπαϊκό PNR. Ή θεωρεί το δικαστήριο ότι αυτό επιτρέπεται γενικώ. Και τέλος, που είναι κάπως υποθετικό, καθότι τοποθετήθηκε το δικαστήριο, εξακολουθώ να μην κατανοώ τα του άρθρου 87 αν δούμε το ιστορικό των συμφωνιών PNR, αρχικά δεν είχαν καμία σχέση με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία, αλλά διαβάζοντας το 87, καταλαβαίνω ότι μιλούμε για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και αντίστοιχη συνεργασία με τρίτες χώρες θεωρητικές απορίες ενδεχομένω γιατί η απόφαση ήταν η απόφαση. Ευχαριστώ Σοφή. Άξελ Φως για το ΕΛΚ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη νομική υπηρεσία για την ανάλυση, τη διεξοδική ανάλυση που παρουσίασε. Καταρχήν να πω πράγματι πολύ καλό αυτό ε, μπορούν ε, να υπάρχουν δυνατότητες ε, να χρησιμοποιεί κανείς το PNR. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν είχα σκεφτεί αυτό το άρθρο 7, την επίκληση του άρθρου 7. Το άρθρο 87 το είπε η Σοφή, το έφυξε αυτό και αυτό πρέπει να σας πω ότι με εξέπληξε λιγάκι. Γι' αυτό θα ήθελα να μας εξηγήσετε λιγάκι Πώς μπορούν να εξηγηθούν όλα αυτά. Πρέπει να σας πω, δεν έχω διαβάσει τη νομική αιτιολόγηση, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω πώς ακριβώς μπορεί να εφαρμοστεί η κοινή νομική βάση και με το άρθρο 87. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι καλό το ότι ε, γνωρίζουμε ότι το PNR πράγματι είναι συμβατό με τη νομοθεσία. Επίσης ε, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι επιτρέπεται αυτή η αποθήκευση δεδομένων μέχρι κάποιο βαθμό βέβαια. Εμείς δεν έχουμε κάνει αυτή τη χρονική διαφοροποίηση που είπατε, δηλαδή πριν από την άφηξη, μετά την άφηξη. Ίσως ε, και εκεί να μπορείτε να με δώσετε περισσότερες πληροφορίες πώς μπορεί να γίνει καλύτερα η εφαρμογή. Όσον αφορά τώρα στα περίφημα ευαίσθητα δεδομένα που θίξατε. Έτσι και αλλιώ τη ρωτάτε κανείς κατά πόσον είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα. Αυτό που με εξέπληξε λιγάκι στην απόφαση είναι ότι στο PNR μπαίνουν μέσα και διατροφικές συνήθειες. Αν δούμε λοιπόν τα δεδομένα και το PNR, το PNR καταρχήν δεν είχε καμία σχέση με τις διατροφικές συνήθειες. Εμένα με εξέπληξε λιγάκι αυτό αλλά πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την απόφαση του δικαστηρίου ήταν ευχάριστο το αποτέλεσμα, δεν ξέραμε καν αν μπορούν να υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες με το PNR. Το Ευρωπαϊκό ε, Σύστημα Προστασίας ε, και το επίπεδο προστασίας ε, κυρίως σε σχέση με τρίτες χώρες Χάρηκα και γι' αυτό όπου υπόθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει, ότι είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η συνεργασία, βέβαια με κάποιο επίπεδο ασφάλειας. Και αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι θα πρέπει ταχύτατα ό,τι δεν γκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να το βελτιώσουμε μέσα από περαιτέρω διαπραγματεύσεις για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει κάποια συμβατότητα. Ακούστηκε ότι η συμφωνία με, την, ε, με τις Ηνωμένες και την Αυστραλία ότι οι συμφωνίε θα πρέπει να, πρέπει να εξεταστούν ενδεχομένως και κάτω από το πρίσμα της πρόσφατης απόφασης. Αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, θα ήθελα να γίνει ταχύτατα, να μην περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Να υπάρξει προσαρμογή σε αυτό που πιστεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά τα άλλα, υπάρχουν και κάποια άλλα ε, κάπως αμεληταία θέματα σε γενικές γραμμές εγώ πιστεύω ότι προχωρήσαμε ένα βήμα περαιτέρω και μπορούμε να δούμε πια τι θα γίνεται με τις μελλοντικές συμφωνίες. Η Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Ε, καταρχήν, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τη νομική υπηρεσία για όλες αυτές ε, τις, τη διεξοδική τοποθέτηση σε αυτά που αποφασίστηκαν από το δικαστήριο. Ε, παλαιότερα πολλοί είχαν ζητήσει απόφαση του δικαστηρίου και εγώ το είχα ζητήσει. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να σας πω ότι σήμερα δεν είμαι ευχαριστημένη. Επιβεβαιώθηκε η θέση μας, αλλά εγώ θα το έβρισκα πολύ καλύτερο το να έχει ασκηθεί κριτική πολύ νωρίτερα και το να είχε προκύψει ένα διαφορετικό κείμενο με βάση αυτά που συζητάμε και σε σχέση με την καλύτερη νομοθεσία, αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο από το να έχουμε μπροστά μας αυτή την τοποθέτηση. Το ότι ε, μπορούν ε, ότι πρέπει να υπάρχει ε, προστασία δεδομένων, αυτό το βρίσκω αυτονόητο. Ας πούμε, σε μία ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν ποσοστά ασφαλείας και σε άλλα όχι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι τα αυτοκίνητα που έρχονται στη δική μου την Ήπειρο θα πρέπει να είναι ασφαλή. Αν λοιπόν αυτό το θέμα μπορεί να γίνεται με τεχνικές διατάξεις, γιατί να μην γίνεται και με την προστασία των δεδομένων. Για μένα όλα αυτά είναι αυτονόητα. Και θέλω να πω και το εξή: Υπάρχει ένα νομικό κενό. Υπάρχει η συμφωνία με τον Καναδά που πρέπει να τύχει επανεπεξεργασίας, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, παρεμφερείς ε, συμφωνίες, μάλιστα με χειρότερες συνθήκες. Και θα πρέπει ως εκ και αυτές να αλλάξουν. Όχι δηλαδή να περιμένουμε να προκύψει μία νέα αγωγή για παράβαση. Εγώ θεωρώ ότι το PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξεταστεί κάτω από αυτό το πρίσμα πριν τελικά εφαρμόζεται. Έχω και μία ερώτηση προς τη νομική υπηρεσία. Αυτή η κατανομή σε διάφορες φάσεις ήταν πολύ χρήσιμη, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Ας υποθέσουμε ότι μαζεύω όλα τα εντομένα και τα διαβιβάζω στην τρίτη χώρα. Και κατά την είσοδο, την άφηξη, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κανένα επικίνδυνο στοιχείο, ούτε και κατά την παραμονή. Κατά την αναχώρηση καταγράφεται ότι δεν υπάρχει τίποτα το επικίνδυνο σε σχέση με αυτό το άτομο, άρα δηλαδή πρέπει να διαγραφούν τα δεδομένα. Και τώρα ερωτώ, ο Καναδάς θα διαγράψει τα στοιχεία που πήρα ή θα τα διαγράψουμε και εμείς, εμείς που τα στείλαμε τα στοιχεία. Ή μήπω είναι αλλιώ, δηλαδή διαγράφει ο Καναδά, αλλά εμεί που τα αποστήλαμε στην αρχή τα διατηρούμε. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστούμε, Birgit. Helge Stevens, παρακαλώ, ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Εμείς πάντοτε υποστηρίζαμε την συμφωνία με τον Καναδά και την αναγκαιότητα της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας για την ασφάλεια των επιβατών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει αναθεωρημένη, επικαιροποιημένη συμφωνία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε με τη συνεργασία μας με τον Καναδά. Ευχαριστώ. Μαρή Κριστίν για την ΚΟΕ θέλατε να επανέλθετε, Σοφή. Μπορείτε αμέσως μετά την επόμενη παρέμβαση. Παρακαλώ. Γιάν Αλμπρεχτ για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την νομική υπηρεσία για την εξήγησή της. Θα συμφωνούσα απολύτως με το ΕΛΚ και το EPR ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να συμμορφωθούμε προς την απόφαση αυτή και να επικαιροποιήσουμε τις συμφωνίες. Και είναι πολύ σημαντικό να μην αρχίσουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγνοούν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το δικαστήριο με την γνωμοδότησή του αυτή, με την απόφαση του αυτή, τοποθετείται επί της συμφωνίας για το PNR και δίδει και την ερμηνεία του για το 8 και το 7 του χάρτη και το 16 της συνθήκης που διέπουν και άλλα μέσα. Υπάρχει λοιπόν μια ερμηνεία της συνθήκης στην απόφαση αυτή η οποία μπορεί να συνοδεύει όλες τις νομοθεσίες, τα νομοθετήματα και τις συμφωνίες μας για να δούμε αν συμμορφούνται και αυτά. Θα ήθελα να εστιαστώ επί του εξής. Η νομική υπηρεσία το είπε ξεκάθαρα και δεν μπορεί να υπάρχει άλλη ερμηνεία ότι δηλαδή το δικαστήριο είπε περαιτέρω τήρηση προσωπικών δεδομένων ανθρώπου ο οποίος δεν θεωρείται ύποπτο ή κίνδυνος σε πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση Τη μεταφορά του ταξιδιού του ανθρώπου αυτού. Αν το δούμε αυτό στα πλαίσια όχι μόνο αυτή τη συμφωνία, αλλά και άλλων και της οδηγία PNR και του κανονισμού εισόδου-εξόδου δεν ξέρω αν είναι κανονισμός ή οδηγία, δεν είμαι σίγουρος εν πάση περιπτώσει εάν ερμηνεύσουμε από κοινού σε όλα αυτά τα πλαίσια που αφορούν στο PNR υπάρχει περίοδος τήρησης και είναι σαφέστατη για όλους αυτούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή, που είναι 4 ή 5 έτη. Και τελικώς δεν υπάρχει καν διάκριση εάν μετά το πέρας περίοδου αυτής είναι ύποπτος ή όχι ο συγκεκριμένος. Επομένως, όλες αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ιδιαίτερα αυτές που, επί των οποίων δεν έχουμε ψηφίσει τελεσίδικα. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ μια συμφωνίας που, είναι, που βασίζεται σε παράνομε διατάξεις. Που δηλαδή τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων μετά το πέρας περιόδου αυτής. Και δεν μπορούμε να ζητούμε από τον Καναδά να είναι πιο αυστηρός με την τήρηση των δικών μας δεδομένων από ότι θα είμαστε εμείς με δεδομένα άλλων υπηκών θα ήταν εντελώς μονομερές αυτό. Το δικαστήριο τοποθετείται γενικώς και στα πλαίσια μιας θεωρητικής ανάλυσης και όχι στα στενά πλαίσια της περίπτωσης της συμφωνίας του Καναδά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς Γιάν. Πρωτού πάω στην Σόφη. Ε, ε, με συγχωρείτε, μία ερώτηση όμως. Να κάνω μία ερώτηση. Γιατί επί τη βάση αυτού που μόλις είπα, θα ήθελα να ρωτήσω την νομική υπηρεσία κατά πόσον θεωρεί ότι θα έπρεπε να συστεθεί να ψηφίσει το Κοινοβούλιο επί του συστήματος εισόδου-εξόδου γνωρίζοντας, έχοντας λάβει υπόψη την αποφασία αυτή του δικαστηρίου. Είναι μια, ένα αδύνατο, μια αδύνατη απάντηση που απευθύνεται μάλλον το ερώτημα προς την νομική υπηρεσία. Ε, πρόεδρε, ένα ερώτημα για τις συνέπειες όλων αυτών πρέπει να επανέλθουμε στη διαπραγμάτευση του Καναδά, στον του δυνατό, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες πολύ λίγο πιθανό μου φαίνεται ότι θα είχαμε ταχεία αναδιαπραγμάτευση υπό την παρούσα διακυβέρνηση. Επομένως, ποια θα ήταν η τελική συνέπεια αν δεν είχαμε επιτυχία αναδιαπραγμάτευσης με χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, στην απόφαση δεν το είδα, αλλά Τι γίνεται με το τυχόν δικαίωμα ενός ενδιαφερομένου να πει ότι ναι, μπορείτε να διαχειριστείτε ή να διαβιβάσετε τα δεδομένα τα δικά μου. Υπάρχει κάποια διασύνδεση απόφασης με τα δικαιώματα των μεμονωμένων πολιτών ακόμα και αν δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο προστασίας να δώσουν την αδειά τους. Σας ευχαριστώ. Κοιτώ και τον χρόνο και θα ήθελα να δώσω στον εκπρόσωπο ε, της υπηρεσίας επαρκή χρόνο. Εν συντομία, για την ίδια την συμφωνία. Ξέρουμε ότι τα δεδομένα μεταφέρονται και την ώρα που μιλάμε συνεχίζουν να μεταφέρονται από τότε που εξέπνευσε η προηγούμενη συμφωνία. Αυτές οι διμερείς συμφωνίες, ό,τι και αν είναι, όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύουν, αλλά είναι και ακόμα χειρότερα γιατί ουσιαστικά συνάδουν ακόμα λιγότερο με τον χάρτη των ε, δικαιωμάτων αυτών. Και ιδιαίτερα μετά τα δικαστική απόφαση. Τι σημαίνει αυτό για τη μεταφορά δεδομένων. Γιατί συνεχίζεται η μεταφορά δεδομένων. Θα προτιμούσα να γίνεται με μια στεναρή νομική βάση. Τι γίνεται με τη μεταμοφορά δεδομένων βάσει εθνικών συμφωνιών. Ευχαριστώ, πολύ. με την υπομονή των διερμηνέων. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 5 και 5. Έχω μία πρόταση. Αν θα μπορούσατε μέσα σε 10 λεπτά να μας απαντήσετε, παρακαλώ. Ελπίζω να είμαι πιο σύντομο, αλλά να προσπαθήσω να σας απαντήσω. Αν τίποτα ξεχάσω να μου το πενθυμίσετε, το ερώτημα του κατά πόσον οι, άντες, οι άλλες συμφωνίες θα εκπνεύσουν αυτομάτως. Είναι ενδιαφέρον να ξεκινήσω με συμφωνίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν συναυτεί. Με το Μεξικό, όπως ξέρετε, βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι σχετικά εύκολο, γιατί θα πρέπει να λεφτούν υπόψη να ουλάσει τα στοιχεία. Η συμφωνία αυτή δεν θα μπορεί να συναυθεί χωρίς να λεφτεί υπόψη το σκέλος αυτό. Άλλες χώρες επηρεάζονται επίσης. Δεν είναι μόνο το θέμα ο Καναδάς, αλλά και το PNR με τρίτες χώρες. Άρα αυτή η συμφωνία δεν έχει ακόμα εγκριθεί και θα πρέπει να δεχθεί υπόψη. Οι υφιστάμενες συμφωνίες είναι δύσκολο. Αναγνωρίζονται από τον νόμο και γι' αυτό λοιπόν όπως εξηγείται το δικαστήριο, με γενναιότερο τρόπο επέτρεψε όλα τα ερωτήματα του Κοινοβουλίου να ληφθούν υπόψη και γιατί κάποια κρατημέλη και κάποια θεσμικά όργανα είχαν αμφισβητήσει καν την παραδεκτότητα της, των ερωτημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δικαστήριο λοιπόν αποφάνθηκε ότι η όλη διαδικασία είχε σκοπό να αποφύγει τις ε, επιπλοκές, γιατί σε διεθνές επίπεδο οι συμφωνίε αυτέ δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι τρίτε χώρε και μπορεί να επιμείνει μία από τα δύο μέρη να εφαρμοστούν. Γιατί στη φάση αυτή λοιπόν δεν θα μπορεί να αποσυρθεί. Δεν θα εκπνεύσουν λοιπόν αυτομάτω αυτέ οι συμφωνίε. Θα παραμείνουν σε ισχύ σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση μόνο σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο με διάφορου τρόπου. με ό,τι προβλέπετε στις ρήτρες της συμφωνίες. Ενδεχόμενη αναστολή, καταγγελία ή ενδεχόμενη ανανέωση. Υπάρχουν λοιπόν μέθοδοι για διαπραγμάτευση ενός τέτοιου σημείου. Αυτό εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο. Η χρηματοδότηση λοιπόν αυτή αφορά μόνο αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία με τον Καναδά, ακόμα και αν ο αντίκτυπο ουσιαστικά ισχύει και σε άλλο. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα συνεχίσουμε και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία. Κατά πόσο όλα τα δεδομένα μπορούν να α, μεταβιβαστούν γιατί πρόκειται για διεθνή συμφωνία. Εν μέρη στέκει αυτό. Νομίζω ότι το δικαστήριο αναφέρεται τη συνθήκη, στη συνθήκη του Σικάγο του 47 που έχει να κάνει με την ε, πολιτική αεροπλοεία και αφορά όλα τα κρατημέλη, όχι όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα. Και βάσει του διεθνούς αυτοδικαίου το δικαστηρίο αποδέχεται ότι όλα τα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν. Αυτό όμως οδηγεί σε ένα ενδιαφέρον ερώτημα κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα για τρίτες χώρες να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό και πώς αυτό θα ίσχυε και θα εφαρμοζόταν στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν ισχύει το διεθνές δίκαιο. Για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ισχύει η σχετική του Σικάγο, τουλάχιστον για τις ε, εισερχόμενες πτήσεις. Αλλά το θέμα θα ήταν πώς θα ίσχυε αυτό και εσωτερικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εσωτερικές πτήσεις, ε, γιατί δεν είναι θέμα διεθνών συνθήκων για την πολιτική αεροπλοεία δεν το αναφέρει αυτό ρητά η γνωμάτευση, αλλά θα πρέπει να το κοιτάξουμε για την νομική βάση τώρα. Ναι. Για την αστυνομική συνεργασία στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το σημείο κίνηση Τα μέρη. Μας ετέθησε γραπτή ερώτηση στην οποία κυκλεθήκαμε να απαντήσουμε. Το δικαστήριο λοιπόν ρώτησε πώς ε, είναι δυνατόν να ισχύει το άρθρο 97 και όλα τα μέρη λοιπόν θα πρέπει να ανταλλάσσουν απόψεις. Υπήρχαν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Το δικαστήριο στην κομματεύση του δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να απαντήσει στην ερώτηση αυτό. Διευκρινίζει ότι ισχύει το άρθρο 97. Αλλά η αιτιολόγηση, να σας πω εμείς μάλλον πώς το παρουσιάσαμε, θα μπορώ να σας το παρουσιάσω από πλευρά ε, Κοινοβουλίου. Υπάρχει ιστορική διάσταση στην αστυνομική συνεργασία, υπάρχει και αντιστοίχως εξωτερική διάσταση όταν η δική μας αστυνομία δηλαδή συνεργάζεται με τρίτες χώρες. Αλλά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί δεν ε, στέλνει η αστυνομία της Ευρώπης ε, στοιχεία στην αστυνομία του Καναδά. Δεν είναι, είναι εμπορική. Οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οντότητες που στέλνουν τα δεδομένα αυτά, υποχρεούνται βέβαια οι εμπορικές εντότητες να στέλνουν τα δεδομένα αυτά. Για το PNR ε, ε θα ε, υποχρεούνταν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εδώ μιλάμε για το καναδέζικο, το καναδικό δίκαιο. Τίφεται λοιπόν το θέμα της αστυνομική εργασίας, ακόμα και αν δεν τίφεται απευθείας αστυνομική εργασία και είναι ενδιαφέρον φυσικά αυτό να το κοιτάξουμε. Και να περάσω στι άλλα ερωτήματα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις άλλες συμφωνίες και να τις ε, επαναδιαπραγματευτούμε. ετέθησε και το ερώτημα του κατά πόσον ο αποστολέας ε, των δεδομένων υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα και αυτό σχετίζεται με αυτό που σας ανέφερα ότι ουσιαστικά οι αερογραμμές είναι αυτές που μεταφέρουν τα δεδομένα σε ό,τι αφορά και το GPTR ε, και το διευκρινίζεται ότι φυλάσσουν τα στοιχεία για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για εμπορικούς σκοπούς θα πρέπει να διαγράφονται σε μετέπειτα χρονική στιγμή και ουσιαστικά επί της αρχής δεν ζητείται, δεν υπάρχει απέτηση να τηρούν τα στοιχεία αυτή. Αντιθέτως θα πρέπει να τα μεταφέρουν παρά αυτά στις αρχές και έτσι λοιπόν η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική. Το ερώτημα του τι συμβαίνει όταν προφανώς δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος και το ζητημα εισοδου εισόδου-εξόδου κυρίως. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Γιατί δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες αυτές, δεν το παρακολουθώ το θέμα, αλλά να απαντήσω επί της αρχής ότι το θέμα επί της αρχής είναι το ίδιο. Αν το αντιστρέψουμε, το θέμα δεν είναι μόνο ότι όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, το δικαστήριο επιμένει μάλλον ότι υπάρχει παρέμβαση σε ό,τι αφορά όταν υπάρχει παρέμβαση στην ειδική σφαίρα θα πρέπει να δικαιολογείται από ενδεχόμενο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πρακτικών στοιχείων που οδηγούν σε υποψία. Θα πρέπει να υπάρχει ρίσκο. Όταν ε, καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ρίσκο, δεν υπάρχει αιτιολόγηση και άρα επί της αρχής όταν διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν δικαιολογείται η διατήρηση των δεδομένων. Αυτό ισχύει επί τη αρχη Για κάθε πράξη τώρα θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι και ποιοι είναι και οι κίνδυνοι πραγματικά. Αλλά αυτό είναι το σημείο εκκίνηση το οποίο αναφέρεται. Θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση βάση κινδύνου και το δικαστήριο επιμένει σαφίστατα σε αποδεντικά στοιχεία, σε αντικειμενικά κριτήρια τα οποία ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ευλογή υποψία. Μία πολύ καλή ερώτηση. Τι συμβαίνει αν οι διαπραγματεύσεις, ε, οι εκ νέων διαπραγματεύσεις δεν πετύχουν, δεν τελεσφορήσουν. Αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο σημαντικό ε, ζήτημα, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς ε, συμφωνία της τρίτης χώρας. Αυτή είναι η θέση η οποία ισχύει για το ευρωπαϊκό δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο ότι αυτά θα περάσουν μόνο αν συμφωνήσει και η τρίτη χώρα σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το δικαστήριο. Αυτό λοιπόν μπορεί να συμβεί μόνο με συμφωνία της τρίτης χώρας. Αν δεν τελεσφορήσουν οι επαναδιαπραγματεύσεις, ποτέ δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί η συμφωνία γιατί δεν υπάρχει τίποτε λιγότερο το οποίο να μπορεί να ισχύσει. Και στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει νομικό κενό και άρα ε, κατά κανόνα επί της αρχής δεν θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρχει νομική συμφωνία, από ουσία νομικής ε, συμφωνίας, διεθνούς συμφωνίας. Θα πρέπει να βρεθεί μια διαφορετική νομική βάση με συνένεση, με συγκατάθεση, ελεύθερη συνένεση της τρίτης χώρας. Αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, θα επικρατήσει μεγάλη επιβολία. Αλλά αυτό που έχει ο Καναδάς κατά τη διάρκεια των δικαστικών αποφάσεων τα τελευταία αυτά χρόνια, τα τρία χρόνια, το Καναδάς υιοθέτησε ένα σύστημα ETS, το οποίο και προτείνει εδώ, όπως και στη ΣΥΠΑ, για να μπορούν να ταξιδεύουν οι επιβάτες στον Καναδά, θα πρέπει να παρέχουν κάποια στοιχεία εκ των προτέρων. Και τέθηκε λοιπόν το ερώτημα του τι θα συμβεί αν τα δεδομένα αυτά χορηγούνται με συγκατάθεση του επιβάτη. Θα χρειαστεί στο μέλλον PNR και ζητήθηκε να απαντηθεί το ερώτημα αυτό γραπτά. Και το δικαστήριο επίσης εξετάσει το θέμα αυτό. Τι θα συμβεί αν υπάρχει συνένεση του επιβάτη. Αυτό επί της αρχής θα πρέπει να υπάρχει ως δυνατότητα τουλάχιστον, αλλά δεν έχουμε τελικά όμως δικαστική απόφαση στο τέλος για το θέμα αυτό. Η συγκατάθεση λοιπόν, εφόσον είναι ελεύθερη, αποτελεί όντως μία δυνατότητα. Ελπίζω να κάλυψα όλα τα ερωτήματα. Αν κάτι ξέχασα, παρακαλώ πείτε μου. Ο Πρόεδρος, συνάδελφοι, συνάδελφοι. Θα σας ευχαριστήσουμε κύριε Μέρφη. Να ευχαριστήσουμε και τα μέλη της Επιτροπής για την γνωμοδοτήση, για την εμπρογνωμοσύνη τους. Να ευχαριστήσουμε και τους εμπρυγνώμονες για την παρουσίαση αυτή. Και να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μέρφ. Τι θα συμβεί αν δεν ε, τελεσφαιρίσουν οι διαπραγματεύσεις, οι νέες διαπραγματεύσεις. Αυτό που πες και εσύ Σοφή. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Συζητούμε και με τη γραμματεία για να είμαστε έτοιμοι και να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό που θα πρότεινα από εσάς θέλω να μου πείτε άμα συμφωνείτε. Πρωτού αρχίσουμε να συζητάμε το κατά πόσο θα τελεσφορήσουν ή όχι διαπραγματεύσει, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι είδου εντολή και η Προεδρία και η Επιτροπή επιθυμούν. Τι προτείνουν πεντολογής. Κύριο Άλμπρεχτ και άλλοι μας ανέφεραν το πώς αυτό σχετίζεται και με τα άλλα μέσα σε ό,τι αφορά το PNR με τον Καναδά, πώς, σε τι σχέση βρίσκεται αυτό με τις δικές μας συμφωνίες με τις αυτές χώρες. Αυτό που προτείνω λοιπόν είναι το, το εξή. Τον Οκτώβριο να καλέσουμε και την Προεδρία, το Συμβουλίο και την Επιτροπή. Είναι και καλή η Προεδρία, είναι η Ιστονή. Μέσα στον Οκτώβριο, γρήγορα για να λάβουμε απαντήσεις. Αν δεν μας δώσουν καλές απαντήσεις για την, ε, το πεδίο της εντολής, φυσικά έχουμε και το ψήφισμα πάντα στο τσεπάκι μας. Αυτό λοιπόν θα ήταν δική μου η πρόταση, να προετοιμαστούμε για μια τέτοια συμφωνία, να είναι συνεκτική, να θέσουμε και αυτά που είπε και ο Γιάνν και οι υπόλοιποι και να προετοιμαστούμε για την ε, συνάντηση, για τη διάσκεψη, για να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Προφανώς από πλευρά περιεχομένου υπάρχει ό,τι χρειάζεται για μια τέτοια προσέγγιση. Αυτό θα μας δώσει λοιπόν και το περιθώριο πρωτοβουλία και ένα δεύτερο σχέδιο, αν θέλετε, ένα plan B για το μέλλον. Αυτό θα μας βοηθούσε, θεωρώ, στο μέλλον. Η Σοφή. Κοιτάξτε, προτείνω. Οι σκιώδεις και εγώ να συναντηθούμε για να ξεκινήσουμε να καταγράφουμε όλες τις ερωτήσεις που έχουμε, να τις στείλουμε στην Επιτροπή σε γραπτή μορφή. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει στο να απαντηθούν οι ερωτήσεις και θα δούμε εάν μετά από μια τέτοια συνάντηση είναι απαραίτητο να υπάρξει ψήφισμα ή όχι. Εγώ θα έλεγα να το έχουμε αυτό κατά νου ότι θα πρέπει να έχουμε εδώ μια πολύ καλά οργανωμένη συνάντηση με την Προεδρία και να τους ρωτήσουμε ποια είναι τα προγράμματά τους. Ίσως ο Γιάνν μπορεί να μας πει τι πιστεύει από αυτού. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι απόψεις είναι πάρα πολύ καλές. Θα ήθελα απλά να ρωτήσω το εξής. Ε, σχετικά με το σύστημα εσόδου-εξόδου πρόκειται να υπάρξει ψηφοφορία και νομίζω ότι είναι καθήκον αυτής της Επιτροπής ε, να επισημάνει στον πρόεδρο ότι εκεί μπορεί να υπάρξει θέμα. Και οι ομάδες και ο Γενικό Γραμματέας πρέπει να συζητήσουν για το θέμα αυτό. Δίκιο έχετε. Μιλάμε για την ψηφοφορία που θα γίνει ήδη τον Οκτώβριο. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσω με τη γραμματεία, να έχουμε μια συνάντηση σαν αυτή που σας ανέφερα πριν από την ψηφοφορία. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε μια ψηφοφορία που να θέτει σε κίνδυνο τη βασική αρχή. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε ε, μια συνάντηση πριν από την ψηφοφορία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε γρήγορα και αυτό σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να έχουμε ένα τέμπο, ένα ρυθμό γρήγορο με τους σκιώδεις. Ξέρω τι έχετε κατά νου. Ότι γίνεται έτσι κάπως ασαφώς λόγο για τη, λόγος για τη συνάντηση, αλλά εγώ ενώ το εξή, εάν υπάρχουν έτσι ασαφείς απαντήσεις, τότε όλα αυτά θα μπουν μέσα στο ψήφισμα. Καταλαβαίνετε φαντάζομαι τι θέλω να πω. Αν θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη πρόταση, να μου το πείτε τώρα. λυπώ που σας εκνευρίζω, λυπάμαι που σας εκνευρίζω λιγάκι. Το θέμα δεν είναι, ε, εδώ δεν πρόκειται για πολιτικά ψηφίσματα. Εδώ είναι το καθήκον μας να εφαρμόζουμε τον νόμο. Και εγώ πιστεύω ότι συνάντηση σκιωδών σε επίπεδο ΛΥΜΠΕ είναι πολύ λίγο για μια επικείμενη ψηφοφορία τον Οκτώβρη που αφορά πολιτικές αποφάσεις της ομάδας αν δηλαδή θα προχωρήσουν στον τριμερή διάλογο και στην ε, πρώτη ανάγνωση. Δεν θέλω ε, μία εβδομάδα πριν ε, να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο. Η Σοφή πρέπει να φύγει πραγματικά και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο το θέμα αυτό και δεν είναι εδώ και ο συγητής. Νομίζω ότι ε, πρέπει να κάνουμε συζήτηση. Η αρχή είναι σωστή. Θα πρέπει να έρθουν εδώ ε, η Γραμματεία του Συμβουλίου, η Επιτροπή. Η αρχή είναι σωστή. Ότι δεν έχει νόημα να πάμε στην ε, Ολομέλεια με ψηφορία και να είναι ανοιχτό το θέμα. Ως εκ τούτου προτείνω να προχωρήσουμε γρήγορα. Και όταν λέω γρήγορα, ενώ αρχές της επόμενης εβδομάδας να βρούμε κάποια λύση. Και θέλω να ε, διατηρήσω την ε, πρότασή μου, ε, να έρθω σε επαφή με το Συμβούλιο, την Επιτροπή και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πριν ε, από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για θέματα εισόδου-εξόδου, για τη σχετική οδηγία. Θα δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Και για το ψήφισμα, ε, παρακαλώ μην το παρεξηγήσετε, είναι ένα πολιτικό όπλο που έχουμε αν δεν μας δώσουν τις ε, επιθυμήσεις, τις απαντήσεις που επιθυμούμε είναι ε, νομικό το όλο θέμα και όχι πολιτικό. Μην παρεξηγήσετε αυτά που λέω. Απλά το λέω για να δω αν έχετε κάποιες καλύτερες προτάσεις. Αν έχετε να μου τις πείτε θα είμαι ευγνώμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη συνάντηση είναι στις 25 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ στην αδελφή όλους. Ευχαριστούμε. The meeting is closed. Λύει τη συνεδρίαση.